Αποχές. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Καταπίπτει 29. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Καταπίπτει και η 31. Είναι ο πρώτος κατάλογο ψηφοφορία που πέφτει στα χέρια μου. Έχετε υπομονή παρακαλώ. Συμβιβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία βρίσκεται μπροστά σας, μπορείτε να τη διαβάσετε λοιπόν. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνατε. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική τροπολογία ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 με την προφορική τροπολογία που μπορείτε να διαβάσετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ας προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξέχασα την κάρτα μου. Δεν την έβαλα στο μηχάνημα. Τι είναι αυτά. Έτοιμοι. Τροπολογία 60. Ψηφίζουμε. 11 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 62. 61, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέραστη της ψηφοφορίας. Δώδεκα υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά απόχέσα. εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε απορρίφθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 16 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 σε δύο τμήμα, ε, τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 19 υπέρ, κατά, αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 20 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία απορρίφθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ε, μία, ε, πρώτη υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Μήπως κάποιος δεν ψήφισε ακόμα. Α, για κοιτάξτε, ισοψηφία απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με τον κανόνα ο κύριος Μαρτά ο κύριος Μαρτά δεν ψήφισε Α, πολύ καλά πολύ καλά τότε απορρίφθηκε ούτως ή άλλως ψηφίζεται υπέρ υπέρ, α υπέρ με συγχωρείτε τότε εγκρίθηκε η τροπολογία. Αυτό δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τις ψηφοφορίες. Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε Πρόεδρε, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Όταν κάποιος λέει ότι δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου, ε, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και το είπε από την αρχή. Ναι, λέει ο κύριο Βίλαντ, αλλά δεν μπορούμε να τον συνυπολογίσουμε. Ναι, το είπε όμως από την αρχή ότι το μηχάνημά του είχε κάποιο πρόβλημα. Εγκρίνεται λοιπόν με μία ψήφο παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να φέρνετε μαζί σας τις ε, κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και να το κάνω κι εγώ επίσης. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου της έκθεσης. Ψήφισαν όλοι, άπαντες, όχι ακόμη. Δύο λείπουν, δύο ψήφοι λείπουν. Κάπου λείπει μία. Πέρα της ψηφοφορίας. 23 και 0 και 3 αποχές. 23 υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές. Πολύ καλά. Κύριε Βαλένθα, σας συγχαίρουμε. Βαλέσα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας μαζί μου. Okay, the people that are leaving the room, please do it now and do it quietly. Όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα, ας φύγουν ήσυχα, ήρεμα, ούτως ώστε να συνεχίσουμε με την εργασία μας. Um, we have you know,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 Έχουμε μια πολύ πλούσια ημερήσια διάταξη, γι' αυτό ας αρχίσουμε. Σας παρακαλώ ε, να κάτσετε στις θέσεις σας, διότι τώρα ε, θα έχουμε την αναφορά ε, για την κοπή της ουράς των χείρων και δίνω τον λόγο στον Οτάβιο Μαζόκη από την, το τμήμα πολιτικής που θα μας κάνει ε, την παρουσίαση. Σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ορών ονομάζομαι Οτάβιο Μαρζόκη από το τμήμα ε, πολιτικής δικαιωμάτων των πολιτών και συνταγματικών υποθέσεων και μας, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια μελέτη που κάναμε κατόπιν ετήσεως ε, της Επιτροπής Αναφορών που έγινε την 1η Απριλίου φέτος που μας ζήτησε να εξετάσουμε το θέμα ε, της αναφοράς για το θέμα της συστηματικής αποκοπής της ουράς των χείρων. Αυτή είναι η δομή της παρουσίασης που θα κάνω. Πρώτα απ' όλα η αναφορά που εξετάζουμε είναι 0336 του 2012 που εξετάστηκε ε, σε δύο, δύο φορές από την Επιτροπή Αναφοράς. Είναι η τρίτη φορά που συζητούμε το θέμα και η συνέχεια που δόθηκε στην Επιτροπή θα εξετάσουμε ε, το θέμα της ε, συστηματικής αποκοπής της ουράς των χείρων σύμφωνα με τον νέο νόμο και μετά θα εξετάσουμε τα μέτρα που η Επιτροπή έχει λάβει για να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας και τα μέτρα που δεν έλαβε η Επιτροπή και που το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει για περαιτέρω μέτρα. Και μετά θα περάσουμε ε, στα συμπεράσματα. Έχετε την μελέτη που διανεμήθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και υπάρχει ένα παράρτημα ε, με τα ερωτήματα τα κοινοβουλευτικά που τέθηκαν στην τελευταία θητεία για το θέμα αυτό και τις απαντήσεις της Επιτροπής. Η αναφορά την οποία εξετάζουμε ε, για την, συστηματική αποκοπή της ουράς των χείρων μας δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη εφαρμογής και παραβίαση της οδηγίας του Συμβουλίου 2008-120 EC που προσθέτει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των χείρων. Υπάρχει ένα παράρτημα σε αυτήν την οδηγία που προβλέπει κανόνες για το θέμα της αποκοπής ουράς των χείρων και ο αναφέρον μας λέει ότι όχι μόνο ε, στην Δανία αλλά και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή και παραβίαση αυτής της οδηγίας. Η Κομισιόν κατά τη διάρκεια των άλλων εξετάσεων στις Επιτροπές δήλωσε ότι ότι ε, δεν κινεί την διαδικασία επί παραβάση εναντίον κρατών μελών, δεν είναι κάτι αποτελεσματικό και η Επιτροπή προσπαθεί να εργαστεί για κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας και να χρησιμοποιήσει μέσα ηλεκτρονικής εκμάθησης και δυνατότητα ενός νέου νόμου πλαισίου για την καλή διαβίωση των ζώων. Η Επιτροπή Αναφορών κράτησε μέχρι σήμερα ανοιχτή την αναφορά, την εξήτασε στις 20 Μαρτίου 2013 και μετά την 1η Απριλίου 2014, οπότε μας ζητήθηκε να κάνουμε μια ανάλυση σχετικά με την αναφορά αυτή και πάλι σήμερα εξετάζεται η αναφορά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να πω, να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με την ορολογία. Τι είναι το ε, δάγκωμα της ουράς. Είναι μια ανώμαλη συμπεριφορά μεταξύ των χείρων που μελετήθηκε από την επιστημονική κοινότητα και η οποία προσδιορίσε ορισμένα στοιχεία κινδύνου ε, και αίτια της, του δαγκώματος όταν ε, οι χείροι βρίσκονται σε περιβάλλον πτωχό που είναι ανιαρό κατά κάποιο τρόπο ή τους προσκαλεί δυσφορία, ε, αυτό είναι το βασικό ε, στοιχείο. Η βασική τους αντίδραση είναι το δάγκωμα των ουρών, δηλαδή ο κάθε χείρος δαγκώνει την ουρά του άλλου. Είναι κάτι το πάρα πολύ σύνηθες σε καταστάσεις όπου υπάρχει ε, ε, εκτροφή εντατική και γι' αυτό η Κομισιό προσπαθεί επίσης ε, να προβλέψει ένα περιβάλλον πιο πλούσιο, πιο εμπλουτισμένο, ούτως ώστε να μην νιώθουν ανία και δυσφορία, διότι η χείρη είναι μεταξύ των πιο περίεργων και έξυπνων ζώων που έχουμε. Επίσης το δάγκωμα αυτό προκαλεί μολύνσεις και επηρεάζει η καλή διαβίωση των χείρων μακροπρόθεσμα και μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες ασθένειες όταν αρχίζουν ε, να δαγκώνουν την ουρά ένας του άλλου. Ε, έχουμε ιούς οι οποίοι ε, μεταδίδονται σε άλλους χείρους. Η συστηματική αποκοπή της ουράς των χείρων, η βασική προληπτική μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους, η συστηματική αφαίρεση ε, μέρους τμήματος ή ολόκληρης της ουράς των χείρων, παίρνουν τα μικρά χειρίδια και ε, χωρίς ε, αναισθησία, χωρίς ε, νάρκωση αφαιρούν την ουρά. Είναι ένας τρόπος πρόληψης του δαγκώματος αλλά δεν επιτρέπει την αποφυγή μολύνσεων. Μπορεί να οδηγήσει χρόνιο πόνο και μολύνσεις και οι χείροι που δεν έχουν πλέον ουρά έχουν μια άλλη συμπεριφορά, δαγκώνουν τα πόδια, δαγκώνουν τα αυτιά. Και μετά, όπως είπαμε, το να εμπλουτίσει κανείς ε, το περιβάλλον τους, ε, το οποίο μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν παραδείγματο χάρη κομπόστα από μανιτάρια, σανό, ψάθα, ε, αυτό θα μπορούσε να μεταβάλει την συμπεριφορά των χείρων και να μειώσει την, ε, το δάγκωμα των ουρών. Η απαγόρευση της ε, συστηματικής αποκοπής φοράς των χείρων περιλαμβάνεται στην οδηγία 2008-120 και υπάρχουν ορισμένοι όροι που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Πρώτα απ' όλα η αποκοπή της σουράς μπορεί να γίνει αν μόνο κοπεί ένα τμήμα της ουράς, δεν μπορεί να γίνεται ε, συστηματικά. Μπορεί να γίνεται μόνο όταν υπάρχει απόδειξη ε, ότι διαδίδεται ή το δάγκωμα το, της ουράς στις εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτρόφοι ε, πρέπει να λάβουν άλλα μέτρα προληπτικά, παραδείγματο χάρη να αλλάξουν τις συνθήκες της περιβαλλοντικές ή το σύστημα διαχείρισης και να λάβουν υπόψη ε, την πυκνότητα των κοπαδιών και το περιβάλλον και ότι η αποκοπή μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο άτομο ή από κτηνίατρο. Θα πρέπει δηλαδή προτού προβεί στην αποκοπή της ουράς ο κτηνοτρόφος να λάβει άλλα μέτρα, να προβλέψει περισσότερο χώρο, παιχνίδια για τους χείρους, υλικό εμπλουτισμού του περιβάλλοντος, να αλλάξει τον εξαρισμό κλπ. κλπ. Επίσης η οδηγία για την οποία μιλούμε είναι 2008, 120 ίση, αλλά έχουμε στον νέο νόμο από το 1991 με προθεσμία, διότι η πρώτη οδηγία που περιλάμβανε την απαγόρευση είναι του 1991, ήταν η οδηγία του Συμβούλου 91-630 EEC αλλά αυτή η οδηγία προέβλεπε μια προθεσμία για τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της μέχρι το 1994. Περάσανε λοιπόν 20 χρόνια από τότε που ο πρώτος νόμος απαγόρευε την συστηματική αποκοπή της ουράς και η κατάσταση είναι αυτή που θα σας παρουσιάσω ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίπεδο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου είναι πολύ περίπλοκο να γίνει κατανοητό διότι η Επιτροπή δεν συνέλεξε συστηματικά πληροφορίες αυτή η ίδια ή τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η απάντηση του Επιτρόπου Μπορτο 2014 τον ε, Μάρτιο σε κοινοβουλευτική ερώτηση όπου λέει σαφώς ότι η Επιτροπή ε, δεν έχει ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον βαθμό ε, τήρησης της απαγόρευσης και ότι ε, οι διατάξεις δεν από την πλειονότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν ξέρει κατά το μάλλον ήτον ότι υπάρχει μια διαδεδομένη παραβίαση της οδηγίας και έλλειψη εφαρμογής, αλλά δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Γι' αυτό αυτό το οποίο κάναμε είναι να εξετάσουμε τις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Έχουμε βάλει εδώ το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ε, της ε, αρχής ε, της ασφάλειας τροφίμων από την Πάρμα το 2007 και τις επισκύψεις που έγιναν από το κτηνιατρικό γραφείο, υπηρεσία που είναι υπηρεσία της Επιτροπής στην DG10 και επίσης μια ΜΚΟ που ονομάζεται Compassionate Farming που κάνει επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις και όπως μπορείτε να δείτε αυτή είναι η συλλογή πληροφοριών ε, και τα κράτη-μέλη, ε, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Λιθουανία και η Σουηδία, τρία κράτη-μέλη από τα 28 τηρούν την οδηγία και σύμφωνα με τις επισκέψεις ε, των υπηρεσιών αυτών. Τέσσερα κράτη-μέλη προσετέθηκαν στις τρεις χώρες, η Κύπρος, η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης άλλες επισκέψεις από την ΜΚΟ Compassioning ε, World Farming οδήγησαν στις, στα ίδια συμπεράσματα. Ε, έχουμε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν τηρούν την ε, εφαρμογή της οδηγίας και προκαλούν ανησυχίες. Είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι υπάρχουν μεταξύ τριών και έξι κρατών μελών που τηρούν την οδηγία ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, παραβιάζουν την οδηγία. Εξετάσαμε μετά τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να ε, προσπαθήσει να βελτιώσει την εφαρμογή. Η Επιτροπή εργάστηκε για κατευθυντήριες γραμμές και για μέσα ηλεκτρονικής εκμάθησης, ενημέρωσης η συζήτηση των κατευθυντήριων γραμμών ε, που υπάρχουν εδώ και δύο χρόνια και έγιναν συζητήσεις, υπάρχουν φήμες σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση είναι πολύ περίπλοκη και επίσης η Κομισιόν ελπίζει να κλείσει, ε, ήλπιζε να κλείσει τη συζήτηση το καλοκαίρι αλλά συνεχίζεται η συζήτηση. Το πρόβλημα με τις κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι δεν είναι δεσμευτικές, δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι συγκεκριμένο αλλά προβλέπουν κάποια καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνουν. Και υπάρχει επίσης και ένα θέμα με την επικοινωνία, διότι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, έχουν εικόνες κλπ. Αλλά είναι κάπως περίπλοκες οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή είναι η εντύπωση που έχουμε. προβλέπουν καθοδήγηση ε, νομική που δεν είναι εύκολα κατανοητή για τον κτηνοτρόφο. Το, ίδιο για τα ε, μέσα, μέσα εκπαίδευσης, εκμάθησης. Ε, είναι δύσκολη η προσβασιμότητα σε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα για τους κτηνοτρόφους. Επίσης, η Κομισιόν χρησιμοποίησε τις επισκέψεις της υπηρεσίας τροφίμων ε, και κτηνιατρικής στα κράτη-μέλη, αλλά δεν είναι μια πραγματική υπηρεσία εποπτείας ή παρακολούθησης. Κάνει ένα πρόχειρη, μια πρόχειρη παρακολούθηση και καμιά φορά ε, αυτή η υπηρεσία όταν ανοιχνεύει μια παραβίαση των απαιτήσεων σε σχέση με την αποκοπή της ουράς κάνει συστάσεις. Άλλες φορές όταν διαπιστώνει παραβίαση δεν κάνει συστάσεις και όταν υπάρχει μια δεύτερη επίσκεψη ελέγχουν και πάλι αν ε, ελέγχουν ή καμιά φορά δεν ελέγχουν αν υπάρχουν περιπτώσεις ε, αποκοπής. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν ο μηχανισμός εποπτείας και παρακολούθησης. Το θέμα της διαδικασίας επί παραβάση είναι κάτι το οποίο το Κοινοβούλιο συζήτησε στις άλλες συναντήσεις με την Κομισιόν στην Επιτροπή Αναφορών και όπως είπαμε η Κομισιόν δεν πιστεύει ότι είναι ε, το πιο αποτελεσματικό μέσο για την τήρηση της οδηγίας. Είναι 20 χρόνια που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και το να έχει κανείς κατευθυντήριες γραμμές 20 χρόνια μετά την απαγόρευση είναι κάτι το πολύ καθυστερημένο. Αυτό θα έπρεπε να το λάβετε υπόψη. Επίσης σε μια κατάσταση όπου βλέπετε ότι υπάρχει συστηματική και επίμονη παραβίαση της οδηγίας. Επίσης η Κομισιό ανέφερε τη δυνατότητα βελτίωσης του νόμου πλαισίου ή να έχει ένα νέο νόμο πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων με δείκτες καλής διαβίωσης, βελτιωμένη εφαρμογή που θα περιλαμβάνει επίσης και το θέμα της συστηματικής αποκοπής της ουράς των χείρων. Αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και θα δούμε τι θα προτείνει η Επιτροπή και η Επιτροπή εργάστηκε επίσης εντατικά για μέσα για την αποφυγή της συστηματικής αποκοπής της ουράς των χείρων. Ελπίζουμε ότι θα έχει ένα υλικό ευχριστό για να αποφεύγεται αυτή η αποκοπή. Τα συμπεράσματα. Όλες οι διαθέσιμες αποδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει υψηλά ποσοστά, ε, συνεχή υψηλά ποσοστά μη τήρησης ε, της οδηγίας από μεγάλη πλειονότητα των ε, κρατών μελών, οι κατευθυντήριες γραμμές, η εκπαίδευση, τα μέσα ηλεκτρονικής εκμάθησης για τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος ε, και εύχριστων υλικών, ίσως ενός νέου νόμου πλαισίου για την καλή διαβίωση των ζώων μπορεί να είναι ε, μέσα τα οποία είναι χρήσιμα. Υπάρχει όμως ε, ανάγκη μιας πιο αυστηρής πολιτικής εφαρμογής, εκτέλεσης οδηγίας μετά από 20 χρόνια απαγόρευσης το θέμα της αποκοπής της ουράς έγινε επίσης θέμα κράτους δικαίου, θέμα ε, υπεροχής ε, του δικαίου, διότι παραβιάζεται ο κανόνας αυτός και κανείς ε, δεν αντιδρά. Υπάρχει δυνατότητα το Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα Ε, το να ε, επισημάνει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη το, το ότι αμελούν να εφαρμόσουν την οδηγία, να χρησιμοποιήσει ένα πολιτικό μέσο εφαρμογής να στείλει η Κομισιόν επιστολή στα κράτη-μέλη για να λάβουν μέτρα και να απειλήσει τα κράτη-μέλη ότι θα κινήσει την διαδικασία επί παραβάση και θα προσφύγει στο δικαστήριο. Υπάρχει ανάγκη συστηματικής συλλογής και ανάγκη να συλλέγονται τα στοιχεία με τρόπο πιο συστηματικό, όπως είπα, να εξασφαλιστεί η εποπτεία και να ε, δημοσιεύονται πληροφορίες για την μεταφορά και τήρηση της οδηγίας, ούτως ώστε το, οι πολίτες να ξέρουν τι συμβαίνει ακριβώς στα κράτη-μέλη και ε, να μπορούν να ασκήσουν τελικά πίεση και θα δείτε στην μελέτη ότι υπάρχει παράρτημα με τα σκηνοβουλευτικά ερωτήματα, ερωτήσεις που τέθηκαν από ευρωβουλευτές από πολλές ομάδες και οι απαντήσεις της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν όλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Οτάβιο. Είναι πραγματικά τεράστιο το έργο σας και βλέπουμε ότι έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Στα συμπεράσματα φαίνεται ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επί τη ευκαιρία είχε αναφερθεί και στη δανέζικη σειρά Μπόργεν. Και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Σουηδία, κανείς δεν έλεγε τίποτα άλλο από αυτό το θέμα της αποκοπής της ουράς των χείρων και πραγματικά υπήρχε έτσι μια αντιπαλότητα Δανίας και Σουηδίας με το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω να δούμε τις λεπτομέρειες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην αναφέρουσα, στους αναφέροντες που είναι μαζί μας ηλεκτρονικά. Η Μπριγκίτε Ντάμ είναι κτηνοτρόφος και σύμβουλος πολιτικής για την εταιρεία Ευημερία των ζώων στη Δανία. waiting for the image Περιμένουμε να έχουμε και εικόνα. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Brigitte Ντάμ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Brigitte Ντάμ. είμαι κτηνοτρόφο και σύμβουλος πολιτικής στην εταιρεία ορθής μεταχείρισης των ζώων της Δανίας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για το ενδιαφέρον που έδειξαν στην αναφορά μας σχετικά με το πρόβλημα της παράνομης συστηματικής αποκοπής της ουράς των χείρων σε όλη σχεδόν την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η τρίτη φορά που απευθυνόμαστε στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Έχουμε ήδη ε, παρουσιάσει το πώς 29 εκατομμύρια ε, χείροι χάνουν πάνω με την ουρά τους κάθε χρόνο στη Δανία και περίπου 200 έω 300 εκατομμύρια χείρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα περισσότερα κράτη-μέλη και σίγουρα στη Δανία αυτή η αποκοπή της ουράς γίνεται συστηματικά χωρίς τις κατάλληλες αλλαγές στη διαδικασία διαχείρισης και το περιβάλλον των χείρων έτσι όπω προβλέπει η οδηγία για του χείρου. Το 99% των χείρων στη Δανία ε, υποβάλλονται αυτή τη διαδικασία αποκοπής της ουράς. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόβλημα αυτό είναι και πρόβλημα της σωστής μεταχείρισης των ζώων και πρόβλημα στρέβλωσης της ε, αγοράς. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα κράτη-μέλη βέβαια που συμμορφώνονται με την οδηγία και αυτό οδηγεί σε μειονεκτική θέση αυτών των χωρών στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι οι χείροι δαγκώνουν τις ουρές των άλλων χείρων ως αντίδραση στο στρες. Καταρχάς χρειάζεται χρειάζονται ε, σωστή, σωστές συνθήκες διαβίωσης και σωστά ε, υλικά ε, εμπλουτισμού για να μπορούν να ε, εμπλουτίζουν και να, να την ε, ζωή τους. Χρειάζονται υλικά για να μπορούν να σκαλίσουν. Και Αυτό όμως δεν είναι μια πρακτική που ακολουθούν οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι και ανταυτού κόβουν τις ουρές των ε, χείρων. Οι χείροι ζουν σε ένα πάρα πολύ στριμωγμένο περιβάλλον, έχουν πάρα πολύ ε, άγχος και αυτό οδηγεί και σε αυτήν την ε, συμπεριφορά. Η έκθεση, η αναφορά μας συγκεντρώνει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την πρακτική αυτή. Υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν στοιχεία που ε, αποδεικνύουν αυτήν την παράβαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από όλα εκτός από έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε συλλέξει και από την κτηνιατρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση της Επιτροπής προτείνει διάφορες λύσεις. Μία από αυτές είναι τα υλικά ηλεκτρονικής μάθησης και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς ε, ε, μπορούμε να ε, οδηγηθούμε στη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη γνώσης, τουλάχιστον όχι στην Δανία ή άλλα κράτη με μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή χείρων. Είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα όπου δεν δίνεται καμία ε, σημασία στις ε, ανάγκες των ε, ζώων, στις βιολογικές ανάγκες των ζώων. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε με το ότι η έκθεση τονίζει την πρόταση να ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα εργαλείο επιβολής της και εφαρμογής της νομοθεσίας ίσως ε, μια πιο σοβαρή αντίδραση να οδηγήσει τα κράτη στο να συμμορφωθούν. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση, διότι αυτή η απαγόρευση ισχύει εδώ και 20 χρόνια και η οδηγία εδώ και 10. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Πέρες Αλβάρες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω. Θα ήθελα να αναφερθώ στην αναφορά και στην έκθεση η αποκοπή της ουράς των χείρων και το πρόβλημα του δαγκώματος στα χειρίδια είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να έχει απλώς μια απαγόρευση. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήθελα να τονίσω. Ε, δεν ε, είναι με μια απλή απαγόρευση και με μια διαδικασία επιπαραβάση που θα λύσουμε το πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε πολύ καλά ότι απαγορεύεται η αποκοπή της ουράς, αλλά θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα καλής διαβίωσης εξίσου σημαντικά, διότι αν σταματήσουμε την αποκοπή θα αρχίσουν τα δαγκώματα ή άλλες συμπεριφοράς που θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Αυτό που θέλω να πω με αυτό είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα απλό πρόβλημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί με μια νομική απόφαση. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω και χρειάζονται πολλές συζητήσεις για να βρεθούν εναλλεκτικές λύσεις σε όλα τα περιβάλλοντα εκτροφίων. Χρειάζονται ειδικά υλικά, εμπλουτισμού, εύκολα εύχρηστα ε, και αλλαγές ε, σημαντικές. Αυτό είναι το τεχνικό πλαίσιο, το γενικό που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι εύκολο να επιληθεί. Σχετικά με τα όσα παρουσιάστηκαν σήμερα, η Κομισιόν σημειώνει την κατάσταση, δεν έχω ε, σχόλια συγκεκριμένα να κάνω. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εφαρμογής της οδηγίας και δεύτερο σημείο επίσης που είναι σημαντικό είναι ότι εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για το θέμα του να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Δεν είναι απλό το θέμα ε, τεχνικό ε, διότι είναι ένα θέμα θεσμικό, όχι μόνο ένα θέμα γεγονότων ε, και υπάρχει διαπραγμάτευση. Όταν υπάρχει μια παράβαση ευρύτατη, σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι εύκολο να επιληθεί γρήγορα. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε λοιπόν για έναν νόμο ε, που θα μπορούσε να υπάρχει στα πλαίσια ενός νόμου πλαισίου. Για την ώρα θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιό ε, έχει μια πρόταση σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και οι προτάσεις παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον εφόσον θα επιτρέψουν να υπάρξουν κέντρα αναφοράς για την καλή διαβίωση των ζώων που δεν υπάρχουν σήμερα και Είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα χάρη στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό που επέτρεψε ε, την ε, ανάπτυξη της επικοινωνίας με τους εκτροφείς. Αν αυτή η επικοινωνία υλοποιηθεί γρήγορα θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στα θέματα επικοινωνίας και ε, εκπαίδευσης, αν θέλετε, κατάρτισης των εκτροφέων για να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την εκτροφή σχετικά με το θέμα ε, της, των μέτρων της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας ε, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η Κομισιό ε, ενδιαφέρεται ε, να εφαρμόζονται καλά οι διατάξεις οι νομικές και αυτό λέχθηκε σαφέστατα από τον, ε, το εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Είναι θέμα δικαίου, θα πρέπει το κράτος δικαίου να είναι σεβαστό. Θα ήθελα να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι τα τελευταία χρόνια ε, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ η Κομισιόν και εργάστηκε για τα θέματα καλής διαβίωσης το 2012 για τις συστοιχίες των οτόκων ορνήθων απαγορεύτηκαν τα κλουβιά ε, ε, και το 2012 και το 2013 μια μεγάλη αλλαγή ε, θεσμική για την διαλογή σε ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Επιτροπή δεν έχει μείνει αδρανής για τα θέματα καλής διαβίωσης αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα υπάρχουν προτεραιότητες και πιστεύω ότι τα κλουβιά σε συστοιχίες είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό η απόφαση που λήφθηκε σε σχέση με το θέμα αυτό και η αλλαγή επίσης είναι σημαντικότητα που έγινε. Το 2014 είχαμε μια σειρά επισκέψεων για το θέμα της σφαγής των νόμων, μια που τέθηκε σε ισχύ το 2013. Τώρα είναι αλήθεια ότι τα θέματα αυτά εφαρμογής έχουν ξεκινήσει καλά και νομίζω ότι η αποκοπή της ουράς θα μπορούσε να περιληφθεί ε, στην ε, ημερήσια διάταξη. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας ε, νέος επίτροπος, μια νέα επιτροπή και τώρα επαναξιολογούνται οι προτεραιότητες. Δεν αποκλείεται το θέμα αυτό που αναφέρετε να ληφθεί υπόψη σε επίπεδο προτεραιότητας αρκετά σημαντικό αυτά και συμφωνώ επίσης για το γεγονός ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μια πολιτική αξιολόγηση κατάστασης ειδική, διότι είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου, γιατί ξέρω πως μας παρακολουθούν στη Δανία. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ε, αναφέροντες, γιατί επέστρεψαν και επέμειναν στην αναφορά τους. Πραγματικά αυτό το θέμα είχε αναφερθεί στην τηλεόραση της ε, Δανίας, η συστηματική αποκοπή της ουράς, των ε, χείρων και η στρεβλώσεις της αγοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την Σουηδία που δεν εφαρμόζει αυτή την πρακτική. Εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό και θα απευθυνθούμε και στην ε, αρμόδια επίτροπο μάλιστα. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι έχουμε παραδεχτεί το γεγονός ότι τα λόμπι έχουν κάνει πάρα πολύ ε, καλή δουλειά. Και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ότι οι καθυστερήσεις είναι φυσιολογικές. Και ότι ο εγκλισμός ε, των χείρων σε αυτούς τους μικρούς χώρους είναι φυσιολογικός. Και ότι αυτό μάλιστα θα βοηθούσε στο να σταματήσει αυτό το δάγκωμα της ουράς. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να ενδιαφέρει ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Δανία υπάρχει μία αντίσταση στην πενικυλίνη σε ορισμένους ε, χείρους και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κτηνοτροφική παραγωγή και, αυτή, και αυτά τα μικρόβια που αντιστέκονται στην πενικυλίνη εξαπλώνονται. Από τη μία λοιπόν παρατηρούμε ότι έχουμε παραμερίσει τελείως οποιουσδήποτε κανόνες ε, ηθικής και ασχολούμαστε μόνο με το κόστος, το οικονομικό κόστος. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση δεν ακολουθείται η αρχή του όποιος μολύνει πληρώνει. Σε αυτή την περίπτωση αυτός που μολύνει, αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση. Δεν είναι μόνο η Δανία βέβαια ε, υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, όπου χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο ε, πενικυλίνη και όπου υπάρχουν πολύ περισσότερα ανθεκτικά μικρόβια. Και αυτά δεν θα... Αυτά τα προβλήματα δεν θα είχαν συμβεί εάν δεν συνέβαινε αυτή η αποκοπή της ουράς στους ε, μικρούς χείρους. Οι καταναλωτές όμως, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία, προτιμούν να επιλέγουν κρέας από χείρους οι οποίοι δεν έχουν υποστεί σε αυτήν την αποκοπή της ουράς και αυτό είναι πιστεύω ένα καλό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε ότι ακόμα ε, ότι μπορείς να πάρεις τους καταναλωτές με το μέρος σου εάν ακολουθείς σωστές ε, κτηνοτροφικές πρακτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συστηματική αποκοπή της ουράς των χείρων είναι κάτι οδυνηρό και πραγματικά βάναυσο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την αναφέρουσα που μας ε, επέστησε την προσοχή και συνεχίζει να το κάνει. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το τι περνάνε αυτά τα ζώα. Η αποκοπή της ουράς είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε. Διότι ακούσαμε και από την αναφέρουσα ότι αυτή η αποκοπή της ουράς γίνεται επειδή δαγκώνουν οι χείροι της ουράς τους. Και αυτό συμβαίνει επειδή ε, υπάρχουν, επειδή ε, ζουν σε άσχημες ε, συνθήκες στις κτηνοτροφικές αυτές μονάδες. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε καταρχάς είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ζώων, να βελτιωθούν οι συνθήκες στους ε, στάβλους αυτούς, οι οποίες είναι πραγματικά παράδεκτες. Αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που θέλουν και τα ίδια τα ζώα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση τα γουρούνια να βρίσκονται κλεισμένα σε ένα στάβλο. Θέλουν να βρίσκονται έξω, να κυλιούνται στη, λάμ, στη λάσπη και να μην δαγκώνουν τις ουρές τους. Όμως δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα κάτω από τις εντατικές ε, συνθήκες κτηνοτροφίας στις οποίες υπόκειται. Η αποκοπή της ουράς δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να αλλάξει το σύστημα. Στις κάτω χώρες υπήρξε μία πρόταση από το κόμμα των ζωόφιλων πρόσφατα να σταματήσει οριστικά η αποκοπή της ουράς των χείρων. Δεν πρέπει πια να θεωρείται το δάγκωμα της ουράς δικαιολογία για την πρακτική αυτή. Και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ότι επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή ένα νόμο πλαίσιο για το θέμα αυτό, ο οποίος είναι κάτι που περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πιστεύω πως πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί με το θέμα της ορθής μεταχείρισης των ζώων, όχι μόνο των χείρων, αλλά και όλων των υπόλοιπων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο για μας, αλλά ακόμα περισσότερο και για τα ίδια τα ζώα. Χρειάζεται επιτέλους εφαρμογή της νομοθεσίας. 20 χρόνια περιμένουμε αυτή την εφαρμογή. Και πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να δώσουμε σε αυτά τα ζώα, σε αυτούς τους χείρους, τη ζωή που τους αξίζει. Χρειάζονται την συμπόνια μας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν συμμορφώνονται ε, με την οδηγία αυτή για την αποκοπή της ε, ουράς και μετά από συστηματικές παραβιάσεις 20 ετών πρέπει πραγματικά η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση. Η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι τα ζώα αισθάνονται και αυτό σημαίνει πως χρειάζονται τη βοήθειά μας. Γι' αυτό λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Θεματοφύλακας των Συνθήκων πρέπει να δείξει αυτήν την συμπόνια στα ζώα παρά να καθυστερεί την διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σημεία. Το ένα, όπως είπε ε, και ο αντιπρόεδρος του Animal Welfare Group ανησυχώ με την ομότητα με την οποία φέρονται πολλοί στα ζώα, στις εκμεταλλεύσεις, στη μεταφορά ε, και στα σφαγεία. Και το πρόβλημα το οποίο συζητούμε σήμερα, η αποκοπή ουρά των χείρων, είναι ακόμα ε, και μια πρόσθετη κατάσταση όπου τα ζώα τους ε, ε, ε, θεωρούνται αντικείμενα και νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να υποστηρίξει οποιαδήποτε αναφορά και ευχαριστώ τον αναφέροντα που, που σχετίζονται με τα ζώα, με την καλή διαβίωση των ζώων. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αποδώσουμε σημασία σε αυτήν ε, την αναφορά και σε οποιαδήποτε άλλη αναφορά αναφέρεται ε, στους φίλους μας που είναι όντα, ζώντα όντα. Το άλλο σημείο είναι ότι το θέμα αυτό υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα για να ρυθμιστεί. Και ε, ανησυχώ για τις συνεχείς παραβιάσεις από τα κράτη-μέλη και δεν έχει γίνει τίποτα για το θέμα αυτό. Είναι ένα γεγονός. 20 χρόνια έχουν περάσει και μόνο τρεις χώρες τηρούν οδηγία. Και ε, Χαίρομαι για τις, τα σχόλια της Επιτροπής ότι δεν είναι εύκολη, εύκολο το θέμα, ναι, αλλά είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα για τους πολίτες μας. Αλλά αν είχε γίνει κάτι στα 20 χρόνια, ε, δεν θα ήταν μόνο τρεις ή έξι χώρες ε, που θα είχαν συμμορφωθεί. Ε, και θα είχαν υποφέρει λιγότερα οι χείροι κατά τη διάρκεια των 20 αυτών ετών. Υπάρχουν τα συμπτώματα, οι αιτίε είναι γνωστές, υπάρχουν οι λύσεις. Τι περιμένουμε λοιπόν, εγώ θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τα σχόλια ε, της Επιτροπής λέγοντας ότι θα επαναξιολογηθούν οι προτεραιότητες, ότι τα ζώα που δεν έχουν φωνή ελπίζω να έχουν προτεραιότητα στην ατζέντα της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κίστερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις. νόημα έχει ένας νόμος που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, καταρχάς. Δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν παίρνουμε αυτόν τον νόμο στα σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να τον εφαρμόσουμε. Και είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν, αν θέλουμε δηλαδή, μπορούμε φυσικά να εφαρμόσουμε τους νόμους μας. Το θέμα είναι ε, πολιτικό. Χρειάζεται πολιτική θέληση. Διότι διαφορετικά βλέπω ότι ή δεν υπάρχει πολιτική θέληση, υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας. Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας μίλησε για αξιολόγηση της κατάστασης. Και πιστεύω πως ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να καλέσουμε τον αρμόδιο επίτροπο. Θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό και πιστεύω πως θα έπρεπε να είχε γίνει και κατά τη ε, διαδικασία για παράδειγμα των ακράσεων. Να ρωτήσουμε τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό το θέμα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και είμαι και ο ίδιος ε, αγρότης και πιστεύω πως ε, πραγματικά όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και ο τρόπος. Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει, τι εφαρμόζεται και τι δεν εφαρμόζεται. Και η οδηγία αναφέρεται σε ε, λόγους όταν υπάρχουν όταν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να αποφευθεί αυτή η αποκοπή της ουράς. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί μια αξιολόγηση της κατάστασης είναι κάτι το πιο γενικό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, πιστεύω πως είτε πρέπει πραγματικά να είμαστε ειλικρινείς και να ακυρώσουμε αυτή την οδηγία, την καταργήσουμε, ή αυτή η αξιολόγηση η οποία αναφέρθηκε να γίνει επιτέλους σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την οδηγία. Διότι βλέπω ότι υπάρχει μια σιωπηλή συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά. Τι θα κάνουμε με αυτήν την αναφορά, θα την αφήσουμε ανοιχτή και μετά όταν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαδικασία επιπαραβάση δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να προχωρήσουμε και είδατε τον κατάλογο με τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται, πόσο μεγάλος είναι, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αποσιώπηση του προβλήματος. Υπάρχουν διοικητικά προβλήματα. Όμως πραγματικά πιστεύω, όπως είπα, ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Ή ας είμαστε ειλικρινείς και ας καταργήσουμε αυτήν την οδηγία ή ας πραγματικά δούμε την κατάσταση ρεαλιστικά, διότι αυτό πρέπει να είναι και το κύριο μέλημα της πολιτικής. Να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε επιτέλους αυτήν την οδηγία. Και εδώ είναι και ένα τυπικό παράδειγμα αυτού που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις να καλούμε τον αρμόδιο επίτροπο για να μας απαντήσει, διότι αυτή η απόφαση είναι και μια πολιτική απόφαση. Θέλουμε δηλαδή ή δεν θέλουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Η κυρία Κόλστα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ δανέζικα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για το ότι έθιξαν το θέμα εκ νέου. Φυσικά και παρακολουθώ το θέμα αυτό στη Δανία και είναι ένα αρκετά ανησυχητικό θέμα. Διότι πραγματικά είναι ανησυχητικό το πόσο συστηματική είναι αυτή η αποκοπή της ουράς των χείρων και το ότι συνεχίζεται αυτή η πρακτική. Είναι ωστόσο περίεργο το ότι θέλουν από τη μία να απαγορευτεί αυτή η αποκοπή της ουράς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το νομικό παραθυράκι που τους επιτρέπει να συνεχίζουν αυτή την πρακτική. Στην ουσία το θέμα εδώ είναι η κτηνοτροφία και έχει να κάνει με χρήματα και πόσα χρήματα εξοικονομούνται με την αποκοπή της ουράς των χείρων. Και εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα ζώα, τα οποία φυσικά έχουν αντίληψη και αισθάνονται και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε. Και εδώ να πω ότι πραγματικά εξεπλάγινα από αυτά που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πραγματικά δεν άκουσα ούτε μία αναφορά σε κάποια δράση που έχει αναλυφθεί δεν άκουσα πραγματικά να λέγεται κάτι, για το ότι έγινε κάτι για την περίπτωση αυτή των χείρων. Έχω ακούσει πολλά να λέγονται για τις, ε, ο, ε, για τις ε, συστοιχίες οτοκίας στα πουλερικά, αλλά τίποτα για τους χείρους. Εγώ στηρίζω, όπως και να έχει, 100% αυτήν την αναφορά και πραγματικά θα με ενδιαφέρει να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελεανόρα έχει το λόγο και μετά θα κλείσω τον κατάλογο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Μάργαρετ, θέλεις και εσύ το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Δεν μπορώ παρά να προσθέσω μόνο όπως ακριβώς το έθεσε και η συνάδελφος μπροστά από μένα το οικονομικό. Εμείς ακολουθούμε κάποια πρότυπα ανάπτυξης, κάποια οικονομικά πρότυπα που έχουν σαν στόχο απλά την ε, ε, οικονομική απόδοση. Οπότε αγνοούμε ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε απαράδεκτα, απίστευτα. Όλοι λοιπόν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, όλοι βρισκόμαστε στην, στο ίδιο μήκος κύματος. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μπροστά μας. Θα πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε πού θέλουμε να προχωρήσουμε και τι πρότυπο ανάπτυξης θέλουμε να ακολουθήσουμε. Διότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης οδηγεί σε τεράστιες ποσότητες επίσης απορριμμάτων και αποβλήτων. Ξέρετε ότι τεράστιες ποσότητες επιπλέον τροφίμων τα οποία προορίζονται μόνο στο να πεταχτούν. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο. Και αν δεν έχουμε εμείς την πρόθεση, την πολιτική να βρούμε κάποιες λύσεις, τότε ποιος θα το κάνει. Τουλάχιστον οι αναφορές μας υπενθυμίζουν ποια είναι τα θέματα πάνω στα οποία πρέπει να εργαστούμε. Σε ευχαριστώ. Μάργαρετ Άουκεν ένα μικρό σχόλιο και τελειώνει η συζήτηση εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μετατρέψουμε το καπιταλιστικό σύστημα και να το μεταρρυθμίσουμε πριν βρούμε μια λύση εδώ. Έχει σημασία να αρχίσουμε να ασχολούμεθα επιτέλους με τις συνθήκες ζωής των ζώων και ιδιαίτερα των κύρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης και το θέμα της υγείας. Γιατί η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι κάποιο πρόβλημα πάρα πολύ, είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, δραματικό θα έλεγα και ένα μεγάλο ποσοστό των ζώων ακριβώς παρουσιάζουν ε, αυτές τις μορφές αντίστασης στα αντιβιωτικά. Πρέπει λοιπόν να μην το αγνοήσουμε αυτό, επιμένοντας στο ότι το κέντρο της προσπάθειάς μας είναι η ευημερία των χείρων. Λοιπόν, ε, αν κατάλαβα καλά, σημειώσαμε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν ένα λεπτομερές ε, σχόλιο για τη μελέτη με πλήρη τεκμηρίωση και αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο δεν έχει ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση βάρος των κρατών μελών. Αν κατάλαβα καλά τα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν ε, μόνο μία προσφυγή τέτοιου είδους στην Γεωργία, στον τομέα της Γεωργίας και αυτό είναι περίεργο. Και γιατί τα κράτη-μέλη να έχουν ε, γενικά την δυνατότητα να παραβιάζουν τον κοινοτικό νόμο, διότι συστηματικά το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι παράλογο, να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ισχύει 20 χρόνια και να αγνοείται η εφαρμογή του. Λοιπόν, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσουν την κατάσταση. Να στείλουμε επίσης τη μελέτη στο Άγκρη και στην Έμβη στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές για να δώσουν αν θέλουν αυτές συνέχεια και σε επίπεδο ευημερία των ζώων και σε επίπεδο γεωργίας γενικότερα. Εφόσον θέλουμε θα μπορούσαμε να θέσουμε επίσης ε, και στις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μας πούν τι δυνατότητες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου, ο οποίος επαναλαμβάνω ισχύει από το 1994 και έχει αποτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει την εφαρμογή του. Θέλετε να συμπεριλάβουμε λοιπόν και την γνώμη των νομικών υπηρεσιών. Καλώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε στο 16 την αναφορά του Μπενεντέτο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Καλαβρία. Είναι εδώ ο κύριος Μπενεντέτο. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο κύριε Μπενεντέτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ και 17 χρόνια η Καλαβρία αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή κατεπίγουσα κατάσταση στον τομέα της, ε, της οικολογίας. Κροτώνε, νότσε, Ούστικα, Ποντιτσέλη, Πιανόπολη, Τζόια, Αντιτάουρο, Τζολί Ρώσο και άλλα μέρα γενικά παράλια και μη αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι ονόματα πόλεων, ονόματα ποταμών φυσικά και αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά σε επίπεδο περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο άπτεται επίσης και της υγείας των πολιτών. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν εκατοντάδες καταχρηστικών... Στα una commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Calabria. Essa ha analizzato le criticità del sistema, ha individuato i soggetti coinvolti είναι σε παράνομες χωματερές αναποτελεσματικές οικονομικά και υπάρχουν και σχέσεις με ε, το οργανωμένο έγκλημα επίσης. Ε, οι υπηρεσίες οι Ιταλικές τα γνωρίζουν όλα αυτά αλλά δεν έχουν αλλάξει τίποτα και η Καλαβρία έχει πραγματικά ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, μόνο 13% διαφοροποιούμενη συλλογή απορριμμάτων. Το κύκλος ε, αντιμετώπισης των αποβλήτων στην ουσία σε ένα μεγάλο ε, βαθμό καταλήγει σε χωματερές παραβιάζοντας και την Ιταλική ε, νομοθεσία που πρόβλεπε ότι το 12 θα έπρεπε να ήμασταν στο 65% της διαφοροποιημένης συλλογής των απορριμμάτων και φυσικά και στην τελική τους κατάληξη που δεν θα έπρεπε να είναι οι χωματερές και οι χωματερές θα έπρεπε να είναι μόνο μια τελευταία αποτάτη λύση. Το σύστημα το διοικητικό της χώρας μου απεδείχθη ανίκανο να μπορέσει να σεβαστεί τους κανόνες και εξόδεψε δύο δις ευρώ με κανένα αποτέλεσμα. Υιοθέτησε αποφάσεις, τις επέβαλε στις τοπικές αρχές χωρίς να αξιολογήσει, να μελετήσει και να διαβουλευθεί ε, παραβιάζοντας τις αρχές της συμφωνίας του άρχους. Συνεπώς λοιπόν το ολοκληρωμένο κύκλο συλλογή των απορρίτων χαρακτηρίστηκε και από έλλειψη προγραμματισμού μέχρι το 2013, από κακή χρήση ποσών, από μη χρήση διαθεσίμων πιστώσεων και από ε, έλλειψη βασικών ε, παρεμβάσεων. Τα δύο τελευταία μόνο χρόνια υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και ε, από απορρίμματα τα οποία σωρεύονταν στους δρόμους των πόλεων αναγκάστηκε να πάρει κατεπήγοντα μέτρα τα οποία αποφάσισε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης που οδήγησε απλά συνολικά τα απορρίμματα αυτά στις χωματερές. Δεν εφαρμόστηκε δηλαδή για μια ακόμη φορά η Ιταλική και κοινοτική νομοθεσία στην Καλαβρία θα πρέπει να υπάρξουν προληπτικά μέτρα για την περισυλλογή ε, των ε, απορριμμάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να ανακυκλωθούν και να ε, αντιμετωπιστούν γενικότερα να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης σεβόμενοι το περιβάλλον και τις νομικές ρυθμίσεις. Η περιφέρεια της Καλαβρίας λοιπόν πρότεινε κάποιες αλλαγές στα πλαίσια του σχεδίου ε, αντιμετώπισης του προβλήματος των απορρίπτων. Αυτό περιλαμβάνει τον στόχο 32,5 διαφοροποιημένη συλλογής ε, απορριμμάτων και όχι 65% το οποίο προεβλέπεται από την Εθνική Νομοθετική Ρύθμιση. Προβλέπεται μια νέα περιφερειακή μορφή οργάνωσης με κόστος το οποίο ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τόνων απορριμμάτων που οδηγούνται σε χωματερές. Αυτό έχει οδηγήσει και σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ε, θα πρέπει να ισχύσει. Διάβασα προσεκτικά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην ε, αναφορά μας. Προβλέπει για το 2014 να κάνει μια ανάλυση σε βάθος του προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων και εκεί όπου ε, φανούν ελλείψεις θα προχωρήσει σε έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε επίσης ότι δημοσίευσε το 2013 και έναν ε, πίνακα δράσης, μέτρων δράσης, που απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας με ορισμένες συστάσεις και λέγοντας ότι μία από τις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές για να μπορέσουν να ζητήσουν οικονομική βοήθεια αφορά τη νομική συμβατότητα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων με το άρθρο 18 της αντίστοιχης οδηγίας του 2001. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και στα πλαίσια του προγράμματος αντιμετώπισης των απορρίτων θα πρέπει όπως είπαμε να είναι συμβατά με το άρθρο 18 της Οδηγίας 28 του 2008. Ε, πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια έρευνα το ταχύτερο δυνατόν να γίνουν τοπικές, ε, ε, τοπικοί έλεγχοι στην Καλαβρία και σε άλλες περιοχές να δημιουργηθεί μια task force η οποία να ερευνήσει, να παρεμβαίνει έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα κρίσιμα επίπεδα στα οποία έχουμε φτάσει τώρα με τα σκουπίδια. Θα πρέπει η Καλαβρία να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο τρόπο προς το όφελος της δημόσιας υγείας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε στην παρούσα φάση. Εάν ναι, παρακαλώ σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη γιατί εγώ μιλάω και σαν πολίτης που έχει υπογράψει την αναφορά αυτή αλλά και σαν ευρωβουλευτής, σαν εκπρόσωπος δηλαδή των πολιτών της Καλαβρίας που ανησυχούν για την υγεία τους και για το περιβάλλον τους. Υπογράψαμε λοιπόν αυτή το, το, αυτή την αναφορά και τη στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί το περιβαλλοντικό θέμα στην Καλαβρία έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι συνέπειες στα θέματα της υγείας είναι τεράστιες. Περιοχές έχουν μολυνθεί, άνω των 700 περιοχών έχει υπάρξει σοβαρή μόλυνση υψηλού κινδύνου και υπάρχουν επίσης και υπεύθυνοι οι οποίοι έχουν προκαλέσει την αύξηση ορισμένων παθολογιών που οδηγούν στην ανάπτυξη όγκων και έχουν θίξει πάρα πολλούς πολίτες της Καλαβρίας και ακόμα και παιδιά χαμηλής ηλικίας. Ε, η λύση των ε, χωματερών δεν είναι σωστή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ανακυκλωθούν, να καλυφθούν και να μην συνεχίσετε να υποβαθμίζετε το έδαφος έχουν υπάρξει θέματα παρέμβασης όπως η εκαθάριση των υδάτων και η χρήση επίσης σαν εναπόθεση επεξεργασμένων αποβλήτων θαλασσίων περιοχών ε, ή και λύσεις οι οποίες έχουν πετύχει σε άλλες περιοχές με συμμετοχή των πολιτών ε, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς ερευνητικούς κύκλους, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος των προτινομένων μέτρων. Εξαρτάται βέβαια από την πολιτική βούληση των περιοχών αυτών. Στα πλαίσια της ε, διακυβέρνησης της περιοχής, της τοπικής, τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν γίνει μέτρα. Θα πρέπει να προωθηθούν μέτρα ανακύκλωσης έτσι ώστε ε, να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση ανακύκλωσης ε, των απορριμμάτων. Ε, θα πρέπει βασικό ρόλο να παίξουν φυσικά και τα κοινοτικά μέσα από το 14 μέχρι το 18 στα πλαίσια της οδηγίας υπαριθμών 98 του 2008. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε το ποσοστό των διαφοροποιούμενων απορριμμάτων, να μειώσουμε τις χωματερές, να υπάρξει μια μεταρρύθμιση ε, του ισχύοντος νομικού πλαισίου, διότι όπως ξέρουμε η διαφοροποιημένη συλλογή απορριμμάτων είναι πολύ πιο χαμηλή από ό,τι προβλέπεται. Με κάποιους λοιπόν συναδέλφους του κινήματος Cinque Stelle έχουμε δημοσιεύσει ένα κείμενο σε σχέση με την κρισιμότητα της κατάστασης στην Καλαβρία. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ή μπορεί να ξεκινήσουν ε, διασώζοντας το περιβάλλον. έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να κάνει μια βάθος ανάλυση και να γίνει αυτό το ταχύτερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία και μια task force η οποία θα μπορέσει να ερευνήσει και να παρεμβαίνει. Έχει τα μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και την δυνατότητα για να διασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή και στην δημόσια υγεία και στην Καλαβριά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαγκανάρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα το πρωί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολήθηκε με μια συγκεκριμένη υπόθεση του 2007 είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις προς το δικαστήριο σε σχέση με τις παράνομες χωματερές της Ιταλίας και της Καλαβρίας φυσικά και καταδικάστηκε η Ιταλία να πληρώσει 40 εκατομμύρια πρόστιμο. Αυτό προστίθεται σε άλλα 42 αναεξάμεινο για τη λειτουργία των παράνομων ε, χωματερών στην χώρα. Αυτό σας το λέω γιατί όπως είναι γνωστό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ενημερώνουμε τακτικά είμαστε εν γνώση της μη κατάλληλης αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων σε όλες περίπου τις Ιταλικές περιοχές. Για την Καλαβρία ειδικότερα τώρα πράγματι είναι μία από τις περιφέρειες της Ιταλίας η οποία προκάλεσε και την απόφαση του δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί στο Λουξεμβούργο για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Από ό,τι φαίνεται στην Καλαβρία υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το 2007. Η οδηγία είναι του 2008 η οδηγία προβλέπει ότι τα προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να γίνονται επίκαιρα σύμφωνα με τις νέες νομικές ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Καλαβρία αλλά και κάποιες άλλες Ιταλικές περιφέρειες. Όπως επίσης και όχι μόνο την Ιταλία αλλά και κάποιες άλλες χώρες. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει κάποιες επίσημες έρευνες και έχει ζητήσει από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και την Ιταλία να δώσουν στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα ενημέρωσης των νομικών ρυθμίσεων. Όλες οι περιφέρειες της Ιταλίας έχουν ενημερωμένα προγράμματα όπως προβλέπει η οδηγία. Ε, συλλέγουμε τις πληροφορίες προς το παρόν και θα πρέπει να ελέγξουμε αν αυτά τα προγράμματα διαχείρισης παρουσιάζουν κάποιες πιθανές ε, ασυμβατότητες με την οδηγία. Η οδηγία δεν καθορίζει ποια είναι τα προγράμματα αυτά, αλλά λέει ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσει στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται για την Καλαβρία για μια ακόμη φορά. Από ό,τι φαίνεται και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους προλαλήσαντες, η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την μεταρρύθμιση του προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας οδηγίας Οι αναφέροντες ε, είπαν ότι δεν φαίνεται ότι έχει υπάρξει διαβούλευση και εμπλακή των πολιτών και του κοινού. Υπάρχει μια οδηγία όμως η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρξει περιβαλλοντικός και στρατηγικός έλεγχος τέτοιου είδους προγραμμάτων. Και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης των προγραμμάτων θα πρέπει να υπάρχει και διαβούλευση με τους πολίτες. Η διαβούλευση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από την αρχή της νομοθετικές διαδικασίες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει το κράτος μέλος για να υιοθετήσει το τελικό σχέδιο. Στην περίπτωση της Ιταλίας υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες είναι υπεύθυνε για την διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων. Οπότε η διαβούλευση ε, στην περίπτωση της Καλαβρίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το, η περιφερειακή κυβέρνηση πάρει απόφαση για να ξεκινήσει η ε, αλλαγή σε επίπεδο νομικό. Υποθέτουμε εμείς ότι όταν το πρόγραμμα αυτό φτάσει σε ένα σχέδιο προχωρημένο και πριν υποβληθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εξετάσει και θα σεβαστεί ε, το τι λέει η οδηγία στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η διαβούλευση με το κοινό και κατάθεση παρατηρήσεων από πλευράς των πολιτών και του κοινού όπως το είπαν και οι προηγούμενοι. Ελπίζουμε ότι αυτό το νέο σχέδιο να δώσει καλύτερα αποτελέσματα, να εφαρμοστεί σωστά και να οδηγήσει σε μια βελτίωση ε, την διαχείριση των αποβλήτων στην Καλαβρία. Τώρα για τους τοπικούς ελέγχους, τον περιβαλλοντικό τομέα, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Εμείς μπορούμε να απευθύνουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη όπως το κάναμε με το roadmap που δημοσιεύσαμε το 2013 για την Ιταλία και για περιφέρειες τις οποίες το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο του Νότου, δηλαδή τις περιφέρειες της Ιταλικές, μεταξύ των οποίων και την Καλαβρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν όπως και στο παρελθόν μπορεί να ξεκινήσει εφόσον χρειάζεται διαδικασίες επί παραβάση για να πιέσει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και αυτό το κάναμε και στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω από τους συναδέλφους πραγματικά να είναι σύντομοι και υπηρεκτικοί. Κύριε Άουκεν έχει το λόγο. Έχουμε πολλές φορές εξετάσει παρόμοια ζητήματα. Πιστεύω πως το θέμα δεν είναι μόνο το ότι κάνει η Κομισιόν με τις ε, δηλώσεις της. Πιστεύω πως υπάρχει ένα μεγάλο βαθύ πρόβλημα διοικητικής ε, φύσης και διαχείρισης στην Ιταλία. Ε, θυμάμαι ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε κάνει μια πρόταση και είχε να συμφωνήσει με 561 διαφορετικούς δημάρχους. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη γραφειοκρατία και πραγματικά πηγαίνεις από τον Άννα στον Καϊάφα. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και ποιος είναι υπεύθυνο και πραγματικά ψάχνω να βρω έτσι λόγια για να το περιγράψω με τον πιο κατάλληλο τρόπο όμως δεν το βρίσκω. Η λύση πιστεύω είναι να ενημερωθούν οι πολίτες και να συμπεριληφθούν στην διαδικασία. Και πραγματικά έχουμε δει ότι ο κόσμος αντιδρά όταν κάποιος κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί θα έχει προχωρήσει πολύ το πρόβλημα. Χρειάζεται επιπλέον και μία συζήτηση μέσα στην Ιταλία για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. διότι αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει πραγματικά να συμπεριλάβει όλους. Αλλά σας παρακαλώ μην ακολουθήσετε το παράδειγμα της Δανίας. Εμείς τα καίμε όλα. Και αυτό οδηγεί σε επικίνδυνες εκπομπές ε, αερίων. Χρειάζεται σύστημα και όχι απλά κάψιμο, όπως κάνουμε εμείς σε όλα. Και πραγματικά όταν άκουσα ότι υπάρχει και στην καμπανία της Ιταλίας έτσι, μια εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων, αυτό με ανησύχησε γιατί μου θύμισε τις δικές μας πρακτικές. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ακολουθήσετε τις σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε, αλλά πραγματικά πρέπει να κάνετε κάτι. Δεν βλέπω κάποιον να ζητά το λόγο. Ο Πέτερ, έχει ζητήσει και εσύ το λόγο. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπω ότι συμβαίνει το αντίθετο από ό,τι με την προηγούμενη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί πραγματικά όλα τα μέσα που διαθέτει για να δώσει μία λύση. Έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάση. Έχουν γίνει δράσεις, έχουν προταθεί λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όμως ε, δεν φτάνουν όλα αυτά. Είναι πολύ καλά αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως χρειάζεται ακόμα περισσότερα. Αυτό που βλέπω να λείπει εδώ είναι η πολιτική θέληση. Και αυτό μου θυμίζει κάποιον που προσπαθεί με γυμνά χέρια να πιάσει ένα ψάρι. Νομίζεις πως το έχεις και μετά σου γλιστράει. Λείπει λοιπόν η πολιτική δύναμη και η πολιτική θέληση στην Ιταλία για να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και το πρόβλημα με τις παράνομες εχωματερές, πραγματικά πιστεύω πως δεν το αντιλαμβανόμαστε σε όλο του το μεγαλείο εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Είναι κάτι που πραγματικά ζητά επίγουσα μεταχείριση και εμείς μπορούμε να λέμε γιατί δεν κάνετε κάτι, όμως σίγουρα δεν είναι και εύκολο φαντάζομαι. Γιατί και να αδειάσουν αυτές οι παράνομες χωματερέ, πρέπει τα απορρίμματα να πάνε κάπου αλλού. Πού θα πάνε και τι θα γίνει στο τέλος. Και αυτή η μεταφορά θέλει χρήματα. Ποιο κερδίζει χρήματα πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να εντοπιστούν οι πραγματικοί αρμόδιοι, οι πραγματικοί υπεύθυνοι και να κληθούν εδώ στις Βρυξέλλες. Πιστεύω. Έχουμε λοιπόν ήδη την διαδικασία επί Έχουμε ε, παγώσει κονδύλια. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και εδώ πραγματικά ακούσαμε διάφορες προτάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία Ένωση 28 χωρών και σίγουρα έχουμε πάρα πολλές ε, πρακτικές τις οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε και από τις οποίες μπορούμε να παραδειγματιστούμε. Ακούστηκε η καύση, ακούστηκε ο διαχωρισμός των απορριμμάτων. Πρώτον λοιπόν ας ακολουθήσουμε, ας δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Δεύτερον ας συνεχίσουμε και ας εντείνουμε τις προσπάθειες που ήδη γίνονται. Και τρίτον ας πραγματικά ψάξουμε να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και φυσικά, όπως υπόθηκε, χρειάζεται να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και τους πολίτες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τόσα χρόνια το συζητάμε και δεν έχει βρεθεί λύση. Η Λεωνόνα έχει το λόγο. Αλλά σας παρακαλώ να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Θα είμαι σύντομη. Να προσθέσω ότι γνωρίζουμε πως ε, τα απορρίμματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απλά σαν απορρίμματα αλλά σαν πόροι, σαν ε, φυσικοί πόροι. Να το υπενθυμίσουμε αυτό και στις Ιταλικές αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση στις εμπλεκόμενες περιφερειακές αρχές της Καλαβρίας ε, λοιπόν, σαν Επιτροπή Αναφορών μπορούμε να αποστείλουμε μία επιστολή στις αρμόδιες περιφερειακές αρχές στην Ιταλία έτσι ώστε ε, να τους προειδοποιήσουμε ε, για να ασχοληθούν σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει μεν στα πλαίσια του πακέτου Waste την, ε, το σύνολο των τρόπων αντιμετώπισης των αποβλήτων ε, αλλά χωρίς να θέλω να μηδενίσω τα πράγματα στην Ιταλία υπάρχουν ε, σε κάποιες περιοχές ε, στο Φριούλ σαν παράδειγμα και στην Κονταρίνα στην βορειοανατολική Ιταλία ποσοστά συλλογής και επεξεργασίας διαφοροποιημένης που ξεπερνούν το 80%. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε στις υπόλοιπες περιοχές της Ιταλίας και της Ευρώπης. Καλώς λοιπόν θα κάνουμε το εξής, θα κρατήσουμε ανοιχτή την οδηγία. Και επίσης βλέπω ότι υπάρχει βούληση της Επιτροπής να εξετάσει ε, το θέμα αυτό ενδελεχώς ε, με βάση την πρόσφατη απόφαση την δικαστική. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εξετάσει, έχει ερευνήσει το θέμα και θα δει λοιπόν η Κομισιόν τι εννοεί ε, το δικαστήριο στην απόφαση του με όλες τις λεπτομέρειες και ίσως μπορεί να θεωρήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Θα πρέπει να ενημερωθούμε περί αυτού. Θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να τηρήσει την δικαστική απόφαση και τις πρόσφατες εξελίξεις. Τι μπορούμε να κάνουμε του χρόνου είναι να ορίσουμε έναν εισηγητή από την Επιτροπή Αναφορών ούτω ώστε να έχει μια θεματική προσέγγιση να εξετάσει τα θέματα αυτά όχι μόνο στην Καλάμπρια αλλά και αλλού. Μια σφαιρική έκθεση, να έχουμε έναν εισηγητή, ένα σκιώδη εισηγητή, οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν πιο συστηματικά πάνω στο θέμα. Μπορούμε αυτό να το πράξουμε. Επιπλέον, όπως η Ελεανόρα επεσήμανε, μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στις αρχές της Καλαβρίας λέγοντας ότι σας παρακολουθούμε, σας παρακολουθούμε σε κάθε βήμα σας, δεν επιτρέπετε αυτό και να τους πούμε ότι η Επιτροπή ΠΕΤΗ παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα ε, και κυρίως ε, για την τήρηση των ευρωπαϊκών διατάξεων. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχετε αντίρρηση? Πολύ καλά. Τότε προχωρούμε. Προχωρούμε τώρα ε, στο θέμα 17 ε, για το τηλεκάνη απορροής του ποτάμου Εύρο. Έχουμε την αναφορά 0938 και έχουμε μαζί μας την Ματίλντα Φοντέν και σας δίνω τον λόγο αμέσως. Θα πάρω το λόγο ε, Εξ ονόματος της κυρίας Μαλτίλντο Ντεφόν. σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε τη δυνατότητα να υπερασπιστώ μια περιοχή ιδιαίτερη και σε επίπεδο περιβάλλοντος αλλά και τόσο εύθραστη όπως το Δέλτα του Έμπρο. Ε, εμείς είμαστε εδώ μια αντιπροσωπεία, έχουμε ετοιμάσει και μια παρουσίαση ε, εκπροσωπούμε κάποιους πολίτες ε, από τις οργανώσεις Τέρες Τελέμπρε. Είμαστε μια οργάνωση εγκάρσια με 40 χρόνια παρελθόν. Εδώ ήρθαμε για πρώτη φορά το 2000 με το Εθνικό Ιδρολογικό Σχέδιο και την ε, μεταφορά της κήτης του Έμπρο στην περιοχή από τον Νότο μέχρι και τη Βαρκελόνη. Εμείς ήρθαμε εδώ να καταγγείλουμε το μη σεβασμό του κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της επεξεργασίας του προγράμματος του ΕΜΠΡΟ. Την τελευταία δέκα ετία έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια σαν εθελοντές για να πάρουμε μέρος σε όλες τις συζητήσεις και τα φόρα και να μπορέσουμε εμείς να επηρεάσουμε προληπτικά και να πείσουμε για το συμφέρον της σωστής εφαρμογής της οδηγίας ε, για τους υδάτινους πόρους και του προγράμματος του υδρολογικού για τον Έμπρο στο μέλλον. Στόχος μας είναι να μην χειροτερεύσει περισσότερο το φυσικό περιβάλλον αλλά από ό,τι φαίνεται ακολουθείται πάντα το ίδιο πρόγραμμα εγκαταστάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων με το παρελθόν και αυτό φυσικά έχει οδηγήσει σε προβλήματα και σε σχέση με την χορήγηση των δικαιωμάτων στο νερό. Ε, έχουν υπάρξει 450.000 νέες άδειες ε, για περιοχές άρδευσης που προστίθενται στις προηγούμενες 965.000. Υπάρχουν επίσης 35 νέοι ε, ταμιευτήρες οι οποίοι προστίθενται στους υπάρχοντες άλλους 44. Ε, οι περιβαλλοντικές μελέτες σχετικά με τη ροή του ποταμού και των παραποτάμων του δεν είναι επαρκής. Ε, το σχέδιο αυτό το οποίο κατατίθεται από πλευράς της, Ιταλικής, της Ισπανικής συγγνώμη, κυβέρνησης είναι παραπλανητικό προϋποθέτει ότι το 75% των υδάτων του ποταμού είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ ο μέσος όρος ο αντίστοιχος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνει το 50%. Αυτό το 75% είναι παράλογο, είναι εκτός πραγματικότητας. Η ανάλυση είναι ατελής και με πάρα πολλές εμπασπεριτώσεις περιπτώσει ε, ε, ελλείψεις. Χρησιμοποιήθηκαν 386 περιπτώσεις ε, ελέγχου από τις 821 στο παρελθόν και ε, φυσικά η ε, στατιστική αυτή είναι ατελής. Χρησιμοποίησαν πάρα πολύ απλοϊκούς περιβαλλοντικούς δείκτες ο ποταμός αυτός και οι ποταμοί μας γενικότερα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να μελετηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Για τη σωστή διαχείριση των υδάτων στην Ισπανία και τη διαχείριση των ποταμών οι ποταμοί αντιμετωπίζονται μεμονωμένοι χωρίς σχέση με, τα, με τις λιβαδικές εκστάσεις τις οποίες διασχίζουν χωρίς να αναφέρεται ότι υπάρχουν ε, ψάρια στους ποταμούς αυτούς και γενικά τους θεωρούν σαν κατασκευάσματα χωρίς ψυχή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σεβαστοί και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν μελετηθεί σε βάθος αλλά το νέο πρόγραμμα, το νέο σχέδιο δεν ε, λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές ε, απαιτήσεις, ιδιαίτερα στα προστατευόμενα μέρη το 75% ε, περνάει μέσα από προστατευόμενες περιοχές και δεν έχουν αξιολογηθεί. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Εμείς καταγγέλουμε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι κάτι το τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τις άδειες για την χρήση των υδάτων. Ε, αυτό ακούγεται περίεργο για τους κατοίκους των βόρειων χωρών της Ευρώπης αλλά για τον Νότο και για τους ε, κατοίκους των περιοχών που διασχίζουν οι ποταμοί αυτοί στον Νότο της Ευρώπης οι άδειε αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, έχει σημασία δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ισπανική κυβέρνηση, θέλει να πωλήσει ουσιαστικά τα δικαιώματα αυτά και στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια νέα προσπάθεια έτσι ώστε να, να μετακινηθεί η κήτη του ποταμού και είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει με απαράδεκτο τρόπο το, ε, το περιβάλλον. Οι περιοχές όπως το δέλτα του ποταμού και οι ευαίσθητες περιοχές, οι χαρακτηρισμένες περιοχές δεν αξιολογούνται ε, και ε, δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις θα έχει η, η νέα προσπάθεια η οποία γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μελέτες ε, οικολογικές έτσι ώστε να μην χειροτερεύσει ακόμα η κατάσταση. Οι προτάσεις που γίνονται και επίπεδο είναι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες ενώ στο παρελθόν οι περιβαλλοντικές μελέτες είχαμε την δυνατότητα να τις εξετάσουμε. Ε, το θέμα είναι βέβαια οι μελέτες αυτές να γίνονται σε σχέση και με τις δυνατότητες μεταφοράς όγκου ε, ε, υδάτων από τον ποταμό όπου αυτό είναι δυνατόν να υπολογιστεί. Υπάρχει μείωση γενικά από ό,τι φαίνεται των υδάτων κατά το 5%. Κατά 5% και για να τα υπολογίσουν αυτά ε, πήραν κάποια σημεία ελέγχου τα οποία είναι εντελώς φανταστικά και εντελώς ε, απαράδεκτα και δεν μπορούν να βοηθήσουν ε, τις καταμετρήσεις γιατί πρόκειται για περιοχές προσκομματικές και δεν έχει υπάρξει κανένα μέτρο για να εξηγήσουν στα ευρωπαϊκά όργανα και στους πολίτες τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της κατάστασης. Υπάρχει επίσης και το θέμα των προσχώσεων. Ξέρετε ότι τα δέλτα δημιουργούνται από τις προσχώσεις τις οποίες προκαλούν οι ποταμοί. Το πρόγραμμα για τον Εύρο αγνοεί εντελώς τα αποτελέσματα, τα αρνητικά που δημιουργούν οι νεοκατασκευασμένοι ταμιευτήρες σε επίπεδο ε, ε, προσχώσεων. Ε, και είναι κάτι το οποίο θα αλλοιώσει την φύση των Δέλτα και υπάρχουν συνέπειες πάρα πολλές αρνητικές εξ αυτού. Συνεπώς λοιπόν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στη μείωση των προσχώσεων. Εν πάση περιπτώσει ε, στην ουσία ε, γίνεται μία προσπάθεια η οποία θέλει να καλύψει τις ελλείψεις και να κάνει το πρόγραμμα αυτό συμβατό με την γενικότερη οδηγία. Έχουν ζητηθεί και πιστώσεις οι οποίες υπολογίζονται γύρω στα 14 εκατομμύρια σε μία πρώτη φάση ε, που θα είναι ένα πάρα πολύ ε, μικρό ποσό το οποίο ε, θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί για 25 χρόνια μετά αλλά στην ουσία θα πρέπει να πληρώσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον με σημερινές τιμές. Ε, νομίζω ότι ποιοι πληρώνουν τελικά όλες αυτές τις υποδομές. Είμαστε εμείς οι πολίτες και φυσικά και γενικότερα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν την οποία θέλουμε να καταγγείλουμε και στο Κοινοβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην οποία καταθέσαμε μία καταγγελία. Εμείς είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς έχουμε τη ζωή μας στις περιοχές αυτές, έχουμε τη δουλειά μας στις περιοχές αυτές ε, και θέλουμε να τα προασπιστούμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε εμείς ε, την, την ζωή μας και τις περιοχές τις οποίες ζούμε. Ήρθαμε λοιπόν εδώ σεβόμενοι τα όργανα τα κοινωνικά για να προστατεύσουμε όπως είπα το μέλλον μας και κυρίως το μέλλον του Δέλτα. Δεν ζητάμε κάτι το περίπλοκο, θέλουμε απλά τον σεβασμό των κανόνων τα, οι οποίοι ισχύουν. Ε, τίθεται να αμφισβητήσει η αξιοπιστία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση του ποταμού Έμπρο. Στόχος μας δεν είναι να καταγγείλουμε οικονομικά, σε οικονομικό επίπεδο τη χώρα μου, όχι σε καμία περίπτωση γιατί αυτό θα μπορούσε να βλάψει τους πολίτες της χώρας μου που ζουν μια οικονομική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά καταστροφική. Εμείς θα θέλαμε το Ισπανικό κράτος να μην συνεχίζει ε, να χρησιμοποιεί με καταχρηστικό τρόπο τα χρήματα των φόρων μας σε έργα φαραωνικά και απαράδεκτα, αδικαιολόγητα. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ληφθούν μέτρα ε, σε σχέση με το ΔΕΛΤΑ τα οποία θα κοστίσουν ακόμα περισσότερο ε, κόστος. Δεν θέλουμε περισσότερο τσιμέντο, δεν θέλουμε περισσότερο μπετόν για την κατασκευή αυτών των νέων φραγμάτων ή ταμιευτήρων όπως θέλετε. Θέλουμε το Ισπανικό κράτος να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει μια λύση να μην ολοκληρωθεί η καταστροφή στα πλαίσια της αναθεώρησης του προγράμματος για τον Εύρωτο το 2015. Εμείς ε, βεβαιώνουμε ότι το νέο σχέδιο από το 15 μέχρι το 21 δεν διαφέρει από το προηγούμενο γιατί είναι κάτι το οποίο αποφασίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι ε, που κάνουν το σχέδιο και για την γενικότερη διαχείριση των υδάτων στην Ισπανία. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχιστούν τα μέτρα τα οποία οδηγούν στην χειροτέρευση και τελικά στην εξαφάνιση του δέλτα του ποταμού. Εμείς σας καλούμε να γνωρίσετε την περιοχή του Εύρω, να γνωρίσετε από πρώτο χέρι όλα αυτά τα οποία σας εξηγήσαμε. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος το οποίο είναι δικό μας αλλά και δικό σας και σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίδεται να υπερασπιστούμε την περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε εδώ, που ταξιδέψατε τέτοια απόσταση για να μας ε, παρουσιάσετε αυτές τις ανησυχίες σας για το περιβάλλον. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αλβαρέγιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, ήδη από το 12 που πήραμε την πρώτη αναφορά είχε ξεκινήσει η εφαρμογή του υδρολογικού σχεδίου και ακριβώς είχαν υπάρξει πάρα πολλές ελλείψεις και για περιοχές της Καταλωνίας και για περιοχές του Νότου. Υπήρξαν, ξέρετε, προσφυγές και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, τον Οκτώβριο ήδη του 2012 καταδίκασε την Ισπανία ε, πιέσαμε λοιπόν για να εγκριθούν τα σχέδια το ταχύτερο δυνατόν. Τον Φεβρουάριο του 2014 έγινε δεκτό το πρώτο ε, σχέδιο για την διαχείριση των υδάτινων πόρων ε, στην Ισπανία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον οποίο κάνουμε και με τις άλλες χώρες σημειώθηκαν πάρα πολλές καθυστερήσεις αλλά όπως είπα αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία έχουμε καταλήξει να τα συζητήσουμε σε επίπεδο διμερές ε, με την χώρα. Αυτό ξεκίνησε τον προηγούμενο Νοέμβριο και θέσαμε στην Ισπανία όλα τα σημεία τα οποία εντοπίσαμε εμείς στα προγράμματα τα οποία εξετάσαμε μέχρι τώρα με στόχο να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των προγραμμάτων τα οποία καλούμεθα να υιοθετήσουμε τον επόμενο χρόνο. Συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες τις οποίες εκφράσατε στο εσωτερικό της αναφοράς σας. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ζητάμε από την Ισπανία εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές των ποταμών της χώρας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Εύρω. είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις ε, στα συστήματα παρακολούθησης ε, και των προσχώσεων, ε, γενικά των περιβαλλοντικών μελετών, τις μελέτες για την χημική οργανοληπτική κατάσταση των υδάτων και των, τις επιπτώσεις σε επίπεδο του υδάτινου ορίζοντα. Γενικότερα για την οικολογική κατάσταση. Αυτές οι δύο κυρίως ελλείψεις τις οποίες προανέφερα οδηγούν στο να χρησιμοποιούνται πάρα, πολλά, πάρα πολλές μάζες νερού οι οποίες δεν έχουν συγκεκριμένη χρήση, δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο. Πολλές φορές περνούν από προστατευόμενες περιοχές και δεν λαμβάνονται υπόψη αυτό. Ε, ε, αντίθετα οι προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να εξετάζονται τακτικά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε αν είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης αυτές οι περιοχές. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι λεγόμενες νέες υποδομές. Είδαμε τα προγράμματα ότι υπάρχει ένα αρκετό υψηλό ποσοστό νέων υποδομών το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί για να, καλυφθούν, ε, ε, να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε υδάτινους σπόρους. Αυτό θα έχει συνέπειες ε, για το σύνολο του νερού το οποίο περνάει από το ποταμό και επίσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με την οδηγία γενικά για τη διαχείριση των υδάτων, την γενικότερη οδηγία όταν δημιουργούνται νέου τύπου υποδομές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή γνώση της οικολογικής κατάστασης των περιοχών αυτών. Λοιπόν αυτά θέσαμε στην Ισπανία μετά από την ανάλυση των προγραμμάτων τα οποία μας κατέθεσε Είχαμε όπως είπα το Νοέμβριο κάποιες διμερείς έπαφες ε, και προσπαθούμε ε, τώρα να ολοκληρώσουμε την έκθεσή μας. Θέλουμε να δημοσιεύσουμε την τελική έκθεση για την αξιολόγηση του Ισπανικού προγράμματος στις αρχές ε, του επομένου έτους, του 2015. Θα υπάρξει μια συνάντηση έτσι και αλλιώς στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Μαρτίου Εκεί θα κάνουμε μια τελική ανάλυση γιατί στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βελτιώσει την κατάσταση αυτή μέσω των μέτρων τα οποία προτείνουμε στις Ισπανικές Αρχές έτσι ώστε ε, και τα επόμενα υδρολογικά προγράμματα τα οποία θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα αποφασιστούν τα επόμενα χρόνια να είναι πλέον συμβατά με τη γενικότερη οδηγία και με τις επιμέρους οδηγίες ε, όπως αυτή για την προστασία της φύσης. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν να ελέγχουμε τη συμβατότητα των ισπανικών μέτρων με τις κοινοτικέ οδηγίες έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε η Ισπανία να εφαρμόσει πλήρως τους στόχους, να φτάσει στους στόχους που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το θέμα και θα δώσω το λόγο στη Σολεδάδ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση που έγινε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αναφέρουσα. Και να ευχαριστήσω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ξεκάθαρα λόγια πάνω στο θέμα και για την αξιολόγηση την οποία έχει κάνει, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται πάντα. Λοιπόν, είναι σημαντικό το θέμα αυτό, ε, το θέμα των υδάτων για την Ισπανία όπως και για το σύνολο ε, του νότου της Ευρώπης. Όπως συνολικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της προστασίας ε, του περιβάλλοντος. Είναι γνωστή η καταδίκη της ε, Ισπανίας για τα προηγούμενα προγράμματα υδρολογικής διαχείρισης τα οποία είχε εφαρμόσει. Ε, γενικά τα προηγούμενα δεν είναι πάρα πολύ θετικά. Και η έλλειψη ευαισθησίας που έχει επιδείξει η παρούσα κυβέρνηση της Ισπανίας είναι κάτι το οποίο δεν μας ε, κάνει παρα πολύ, μα πολύ επιφυλακτικούς. Χαίρομαι λοιπόν γιατί είναι σημαντικό να δημοσιευθεί και αυτά, να δημοσιευθούν τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από τις διμερείς επαφές και καλό θα ήταν να γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία τα οποία ανέφερε η Ισπανική πλευρά στα πλαίσια της διμερούς αυτής επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για το αν είναι δυνατόν να κάνουμε μία επίσκεψη ή όχι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να συνεχίσουμε εν πάση περιπτώσει να παρακολουθούμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και να δούμε ακριβώς και ποια θα είναι η πορεία την οποία θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της αξιολόγησης σε έφθετο χρόνο των μέτρων αυτών. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί και θα ήθελα κάπως πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους από την Οργάνωση Προστασίας του Περιβάλλοντος που ήρθαν εδώ για να προασπιστούν το περιβάλλον μας και να προασπιστούν κάτι που όλοι επιθυμούμε. Πράγματι Υπάρχει μια οδηγία η οποία έχει εφαρμοστεί και στα πλαίσια της προστασίας άλλων παραποτάμιων περιοχών της Ιταλίας, της Ισπανίας, συγγνώμη, όπως αυτή του ποταμού Τάγου κτλ. Υπήρξαν και άλλες αναφορές λοιπόν οι οποίες είχαν γίνει δεκτές στο παρελθόν αν και δυστυχώς δεν έχουν μέχρι τώρα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Για την συγκεκριμένη οδηγία αναφερόμαστε λοιπόν για την περιοχή του Δέλτα του Εύρου και της περιοχής γύρω από το ποτάμι του Εύρου γιατί δυστυχώς τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα απολύτως ε, αρνητικά για το περιβάλλον και την κατάσταση του ποταμού, ήταν ε, αρνητικά επίσης γιατί ε, ελήφθησαν για να εξυπηρετήσουν ανάγκες οι οποίες ήταν εις βάρος της φύσης ε, και δεν είχαν καμία ουσιαστική κοινωνική χρησιμότητα. Ε, και αν υπάρξουν ε, περαιτέρω κατασκευές νέων ταμιευτήρων, νέων μικρών φραγμάτων για την ε, διεύρυνση των περιοχών ίδρευσης γύρω από το ποτάμι, αυτό θα προκαλέσει πολύ περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα και θα είναι φυσικά ένδειξη μη εφαρμογής των αρμόδιων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μη σεβασμό γενικά των μέτρων για το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε εμείς να υπάρξει μια αποστολή έρευνας στην περιοχή αυτή. Ξέρουμε επίσης ε, ότι υπάρχουν ε, στα πλαίσια της Natura 2000 στην περιοχή αυτή εκατοντάδες σημεία και μέτρα ενδιαφέροντος ε, τα οποία έχουν σχέση άμεση με την προστασία του ποταμού και γι' αυτό ακούσαμε με ενδιαφέρον αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές παραποτάμιες και όχι μόνο στον Εύρο. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το σχέδιο το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές οδηγίες έγινε πρόσφατα δεκτό όταν ο κύριος Κανιέτε ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος και τώρα που είναι επίτροπος ίσως τελικά να μπορέσει να φανεί και χρήσιμος. Thank you. Mr. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος. Θα ήθελα και εξ ονόματος των Πρασίνων να ευχαριστήσω ε, για την παρουσία τους εδώ και την υπομονή τους της εκπροσώπους της, ε, του Συλλόγου Προστασίας του Ποταμού. Γιατί ξέρω ότι έχουν έρθει πολλές φορές εδώ και ασχολούνται με πάρα πολλά χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά μια προστατευόμενη αν πολύ σε περιοχή μας έχει απασχολήσει όπως είπα και δείχνει ότι η κυβέρνηση ε, του ε, ε, Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία αγνοεί τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των υδάτων και το θέμα των υποδομών τις οποίες προγραμματίζει είναι κάτι το οποίο μας κάνει καχύποπτους ότι το νέο αυτό υδρολογικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και κάτι το οποίο δεν επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι απαραίτητο. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα να ζητήσω όπως η κυρία Ομπιόλ να δημιουργήσουμε μια επιτροπή έρευνας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πόσο μπαίνει προς τα μέσα στην υπηρετική χώρα πλέον το θαλάσσιο νερό σε μια κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική. Πρέπει σαν Επιτροπή να το δούμε αυτό για να πιστούμε. Να ζητήσω επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και προσεκτική στα θέματα αυτά γιατί σε ό,τι αφορά το περιβάλλον είδαμε ότι υπάρχει μια κακώς εννοούμενη ευελιξία στα πλαίσια της ανάλυσης η οποία έχει γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή εφαρμογή μια αυστηρή εφαρμογή των ε, κανόνων που είναι σε ισχύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους αναφέροντες εκ μέρους του ΕΛΚ. Πραγματικά παρατηρήθηκε κάποια καθυστέρηση από πλευράς της ε, προηγούμενης σοσιαλιστικής κυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και αυτό, αυτό το αυτό φάνηκε και από, το, από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2014. Το σχέδιο για τον ποταμό Εύρω έχει επιπτώσεις και στην, ε, στην αυτονομική ενότητα της περιοχής. Εγκρίθηκε με 72 ψήφους υπέρ και 9 κατά το σχέδιο αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί. Αυτό που πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε την ε, τελική και οριστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα Έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την έκθεση στις αρχές του επόμενου έτους και εκεί θα δούμε αν η κυβέρνηση της Ισπανίας έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως πρέπει να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να περιμένουμε την τελική έκθεση. Και δεν πιστεύω πως χρειάζεται διερευνητική αποστολή από την Επίτροπή μας για να δούμε εάν έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά μέτρα. Δεν θα πρέπει, πιστεύω, να παρέμβουμε στη διαδικασία, προτού γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι συμβαίνει. Και πραγματικά να δούμε εάν όντω υπάρχουν θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και μετά να τα επανεξετάσουμε. Έτσι πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσουμε. Η Μπεατρίς, ευχαριστώ. Θα ήθελα εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω τους, τις αναφέρουσες για την παρουσία τους εδώ. Είναι πράγματι η ανάγκη να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν όπως είπατε και εσείς. Καταρχάς σε σχέση με την ενημέρωση που μας έκανε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις τις οποίες παρουσιάζει το συγκεκριμένο σχέδιο. και να συμπεριληφθούν οι ελλείψεις αυτές στην τελική έκθεση την οποία θα συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει με ξεκάθαρο τρόπο ε, να κάνει τη δουλειά αυτή σε επίπεδο ε, υψηλό λεπτομέρειας. θα πρέπει να είναι κατανοητές οι παρατηρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενημερωθούμε σωστά. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας έτσι ώστε να μας παρουσιάσει το σύνολο των ελήψεων αυτών του προγράμματος του Ισπανικού. Σχετικά τώρα με την πιθανή επίσκεψη, την ερευνητική, εμείς έχουμε κάποιους κανόνες ε, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας μας και θα πρέπει φυσικά να σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς. Ε, μια μελέτη ε, πρέπει να έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο και τη συνάντηση με πολύ συγκεκριμένους εμπλεκομένους και έτσι θα γίνεται μια τέτοια επίσκεψη, αλλά θα πρέπει αυτό να το συζητήσουμε εκ των προτέρων σε επίπεδο συντονιστών. Τώρα το να συζητήσουμε τώρα το θέμα της πιθανής επίσκεψης είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει την παρούσα στιγμή. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε εξαιρέσεις εκτός και αν οι συντονιστές αποφασίσουν ότι υπάρχουν τα επαρκή στοιχεία το οποίο θα τεκμηριώσουν τη συγκεκριμένη εξαίρεση. Λοιπόν, ε, θα πρέπει ίσως σε έκτακτη φάση ε, ε, να προβλέψουμε μια τέτοια επίσκεψη, εφόσον βέβαια λάβουμε και την ενημερωμένη πλέον έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι ο λόγος που συζητούμε αυτή την αναφορά σήμερα είναι ότι θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών πού θα πάμε για αυτές τις επισκέψεις μελέτης δεν μπορούμε να λάβουμε μία απόφαση για μια τέτοια επίσκεψη προτού εξετάσουμε διεξοδικά τη σχετική αναφορά και γι' αυτό το συζητάμε σήμερα. Τώρα το λόγο έχει η Άστερ Εράντς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής σας εγώ δεν είμαι τακτικό μέλος, αλλά ενδιαφέρομαι για τα θέμα αυτό. Ε, πρώτον, ε, γιατί επαγγελματικά ασχολούμαι με τα θέματα του περιβάλλοντος και δεύτερον, προέρχομαι από την συγκεκριμένη αυτή περιοχή από τη, γύρω από τον ποταμό. Και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τις αναφέρουσες και για την παρουσία τους εδώ και νομίζω ότι αντιμετωπίζουν το θέμα με σωστό τρόπο. Άκουσα επίσης και είναι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των διμερών επαφών. Ήταν μια καλή ευκαιρία γιατί είδαμε τι λεπτομέρειες μπορεί να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από τα θέματα που αφορούν την ε, περιοχή του ποταμού Εύρω. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και μέσα από τις επαφές αυτές να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να δίδει εγγυήσει ε, στους πολίτες. Συνεπώς λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν κυβέρνηση εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ισπανική κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα αν υπάρξουν πιθανές ελλείψεις και έλλειψεις, ελλείψεις συμβατότητας πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα στοιχεία αυτά στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα περιμένουμε λοιπόν να εντοπιστούν τα σημεία αυτά, τα προβληματικά σε σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Ισπανικό κράτος έχει επιδείξει μια πλήρη αποφασιστικότητα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και νομίζω ότι θα βρεθεί ε, μια κάποια λύση. Τώρα δεν τίθεται το θέμα της παρακολούθησης των μέτρων εφόσον ακόμα δεν έχουν οριστεί σωστά. Λοιπόν, και οι εκπρόσωποι της Ισπανικής Δημόσιας Διοίκησης και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι μπορούν να μας ενημερώσουν σωστά. Από τον Επίτροπο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο είναι ικανοί να παρακολουθήσουν το θέμα αυτό και να μας ενημερώσουν σωστά. Δεν ξέρω γιατί ε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι απόντες, αλλά νομίζω ότι οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το θέμα αυτό είναι σε θέση να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους ε, με σωστό τρόπο. Λοιπόν, εγώ όπως σας είπα προέρχομαι από την περιοχή του ποταμού ε, εγώ επίσης ε, γνωρίζω πολύ καλά και λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης σε τα θέματα του περιβάλλοντος και τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τίθενται σε σχέση και με το Δέλτα του ποταμού και υπάρχουν πάρα πολλοί παραπόταμοι οι οποίοι ε, ε, ποτίζουν περιοχές της Ισπανίας πολύ μακριά από τον ε, ποταμό, από το κύριο σώμα του ποταμού. Λοιπόν, πρέπει να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες του ποταμού και σε σχέση με τις ρυθμίσεις γύρω από τις παραποτάμιες περιοχές. Στην περιοχή της Αραγών, σαν παράδειγμα, τα προγράμματα είναι ατελή ενώ το νερό του ποταμού είναι απαραίτητο για να επιβιώσει η περιοχή. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν ρυθμίσεις έτσι ώστε και οι αρχές σε επίπεδο προστασίας οικολογικής να γίνουν σεβαστές και οι περιοχές γύρω από το ποτάμι να μπορέσουν να επιβιώσουν. Thank Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους ευρωβουλευτές στον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε όμως μία ακόμα αναφορά να εξετάσουμε σήμερα και από ό,τι κατάλαβα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μείνει ανοιχτή η αναφορά για περαιτέρω διερεύνηση από εμάς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε την ε, συμμόρφωση και την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Αυτή η οδηγία πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω και θα περιμένουμε λοιπόν αυτή την αξιολόγηση. Θα περιμένουμε επίσης και τα αποτελέσματα του διαλόγου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κυβέρνησης της Ισπανίας. Και έτσι λοιπόν θα πράξουμε και στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητήσουμε την αποστολή αυτή μαζί με τις υπόλοιπες ε, διερευνητικές αποστολές που έχουν προταθεί. Αυτά για σήμερα προς το παρόν. Συμφωνείτε με την διαδικασία. Θεωρώ πως συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο και τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης, η αναφορά 1957 του 2012 από τον Μαριάνο Βελάσκο Λισκάνο για την διαχείριση του υδρολογικού σχεδίου της περιοχής Άλτο Γκουαντιάνα. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με την συγκεκριμένη οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση αναλύει τις πληροφορίες τις οποίες έχει αποστείλει ο αναφέρον. Η γνώμη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα σας μεταφέρουμε είναι ότι η ολοκλήρωση του άρθρου 6 του προγράμματος του υδρολογικού για την Άλτα Γουαρδιάνα δεν είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με το κοινοτικό κεκτημένο. Ανεξαρτήτως όμως των μέσων που θα θέσει σε εφαρμογή ένα κράτος μέλος, στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να τηρηθούν ε, οι διαδικασίες επίτευξης των στόχων της οδηγίας κάθε φορά. Λοιπόν, η ουσία του προβλήματος μας απασχολεί, μας απασχολεί επίσης ε, η υπερεκμετάλλευση των πόρων της περιοχής. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία έχω πει. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε και στο Νοέμβριο στα πλαίσια της διμερούς επικοινωνίας εμείς ζητήσαμε να υπάρξουν οι κατάλληλοι έλεγχοι έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις ποσότητες των υδάτων οι οποίες αφαιρούνται από την ροή του ποταμού και να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα των υδάτιμων πόρων και ιδιαίτερα για ιδιαίτερα εμβληματικές περιοχές υψηλής προστασίας Εν πάση περιπτώσει μας απασχολεί ιδιαίτερα ε, η διαχείριση των υδάτων στη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι η αρχή της πρόληψης ε, που περιλαμβάνεται στη συνθήκη πρέπει να εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. <coughs> Λοιπόν, η λογική την οποία χρησιμοποιούμε ε, στα πλαίσια αυτού του θέματος είναι η ίδια που χρησιμοποιούμε και στην προηγούμενη περίπτωση και ελπίζουμε να μπορέσουμε στις αρχές του επόμενου χρόνου να δημοσιεύσουμε την τελευταία μας μελέτη, την τελική μας μελέτη για να υπάρξει μια σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τα, ε, ε, για τα ύβατα. Ευχαριστώ. Thank you. I have Soledad. Ευχαριστώ πολύ. Η Σολεδάδ έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ασχολούμαστε πάλι λοιπόν με αυτό το θέμα που αφορά την οδηγία πλαίσια για τα ήθατα και πάλι πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση της Κομισιόν και να την λάβουμε υπόψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει μια τέτοια αξιολόγηση από την οποία μπορούμε να εξάγουμε πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Και πρέπει επίσης να πληροφορηθούμε περισσότερα για την διμερή συνάντηση Επιτροπής και ε, Ισπανικής Κυβέρνησης. Η κυρία, κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε σε επαφή με τον αναφέροντα, ο οποίος μας είπε ότι δεν ήξερε ότι η αναφορά του επρόκειτο να εξεταστεί εδώ σήμερα δεν ήξερε ούτε καν ότι η αναφορά του είχε μείνει ανοιχτή. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία νομίζω. Ε, δεν ξέρουμε ποιος φταίει, αλλά κάποιος θα φταίει νομίζω. Ο αναφέρον μας λέει ότι το 2013 το υδρολογικό σχέδιο της περιοχής Γκουαντάνια υιοθετήθηκε και κατά αυτόν Υπάρχει πολλαπλασιασμός επί 2 ή επί 3 της εισφοράς από τους σπόρους, κυρίως με την περιοχή Μοντιέλο για, κατά το γνώμη του δεν υπάρχει τήρηση της οδηγίας πλαισίου. Ε, το, η υπολεκάνη της περιοχής Αλτο Γκουαντάνια κινδυνεύει κατά τη γνώμη του και μας εξηγεί τον αντίκτυπο ε, επιδίνωσης πάνω σε αυτήν ε, την, την υδάτινη υπόγεια μάζα η οποία είναι σε κακή ε, χημική κατάσταση με λόγω των θιούχων και δεν υπάρχει κανένα μέτρο για την μείωση αυτού του αντικτύπου. Για να τηρηθεί λοιπόν η οδηγία πλαίσιο υιοθετήθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα παρά την ύπαρξη εφαρμογής του σχεδίου αυτού εφόσον το κονσόρσιουμ για το ειδικό αυτό σχέδιο διαλύθηκε και de jure η οδηγία πλαίσιο για το είδωρο δεν τηρείται στο, στην περιοχή Αλτογκουαντάνια. Αυτό μας λέει ο αναφέρον και αυτό ήθελα να προσθέσω απευθυνόμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε λοιπόν να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά περιμένοντας την αξιολόγηση της Επιτροπής Ο αναφέρον μας επεσήμανε ότι θα μας μεταδώσει νέες πληροφορίες και νέα στοιχεία που δείχνουν ε, την μη τήρηση της οδηγίας πλαίσιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια περίπτωση παρόμοια με την προηγούμενη ο αναφέρον ε, μας λέει ότι η διάλυση του κονσόρσιουμ είναι ε, παραβίαση της οδηγίας ε, πλαισίου, διότι κάθε ε, κράτος μέλος θα πρέπει να έχει μια διαχειριστική αρχή και η διάλυση του κονσορσίου μας δείχνει ότι δεν υπάρχει τήρηση της νομοθεσίας εφόσον τα μέλη του κονσόρσιουμ, δηλαδή το κράτος και η περιοχή Καστήλης Μάντσα, δεν, έχουν διαλύσει αυτό το consortium. Η Κομισιό αναλύει αυτήν την έκθεση. Ας περιμένουμε την έκθεση και την αξιολόγηση της Κομισιό και μετά θα αποφανθούμε και θα δούμε αν σύμφωνα με την Κομισιό ε, υπάρχει αυτή η παραβίαση της νομοθεσίας. Ο καθένας κάνει την ε, δική του αξιολόγηση Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να ακούσαμε τι είπε η Κομισιό. Νομίζω ότι βεβαίω οι πολιτικοί δεν ξέρουν την απάντηση. Περιμένουμε την έκθεση της Κομισιόν. Δεν έχω άλλον που να θέλει να λάβει τον λόγο. Ας κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν αναμένοντας τα συμπεράσματα της Επιτροπής σε αυτήν την περίπτωση ε, ε, θα δούμε αν έχει ενημερωθεί ο αναφέρον, ο αναφέρον έχει τις ίδιες πληροφορίες και πρόσκληση για συμμετοχή ταυτάχρονα όπως και άλλοι αναφέροντες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ενημερώθηκε αλλά περιμένουμε ούτως ή άλλως τις πρόσθετες πληροφορίες, αλλά προσεκλήθη την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα όπως και άλλοι αναφέροντες. Αυτό θα πράξουμε και θα ζητήσουμε από την Κομισιό να επανέλθει με τις τελικές πληροφορίες. Νομίζω ότι θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό γεύμα, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, έχουμε την ακρόαση σήμερα το απόγευμα στις 3 η ώρα. Στις 3 η ώρα. Θα βρεθούμε στις 3 ε, η ώρα. Ναι. Έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε έναν κατάλογο εδώ με αναφορές. Λάβαμε πληροφορίες με email, έχουμε πληροφορίες για τον κατάλογο και συμπεραίνουμε λοιπόν σας εύχομαι ε, καλό γεύμα και θα βρεθούμε αργότερα.